Ψηφίζουμε λοιπόν. Θα πάμε με τη σειρά. Πρώτα, η κυρία Φράνσις Ρουάν. Φράνσις Ρουάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία πάλι. Πέρας. 23 υπέρ, 5 κατά, 5 εποχές. Εγκρίνεται υποψήφια. Δεύτερος, ο κύριος Κάι Κάρτενσεν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 26 υπέρ, 5 κατά 2 εποχές. Και τώρα η κυρία Μιρέγ Ελμπάουμ ή Ελμπόμ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 25 υπέρ, 3 κατά, 6 εποχές. Όλοι οι υποψήφοι εγκρίθηκαν. Συγχαρητήρια σε όλους τους ολοκληρώνουμε αυτή τη σύντομη ψηφοφορία. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι ακριβώ ε, η εξέταση των ε, τεχνικών προδιαγραφών για την αποτίμηση για στόχους εξυγίανσης ε, και οι διαφορές ε, της εξυγίανσης υπό το καθεστώς BRRD. Και αυτά είναι στο άρθρο 36 και 74 του σχετικού κανονισμού. και βασιζόμαστε στο κείμενο που μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή τον Μάιο του 2017 θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον κύριο Μιλιάνο Τουρνέζε από τη Γενική Διεθνής Φίσμπα και τον Σπυρίδωνα Ζάρκο από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Δεν έχουν έρθει. Α, δεν έχουν μπει μέσα. Μάλιστα. Χρειαζόμαστε δύο λεπτά για να περάσουμε μέσα γιατί ήμασταν σε συνεδρία κυκλισμένων των θυρών. Θα σας διασκεδάσω εγώ λοιπόν, περιμένοντας. Δεν ξέρω, μπορείτε να δείτε αν οι κύριοι Τουρνέζη και Τσάκος είναι εδώ. Okay, I can give you some background also to underline uh, area where some member expressed some concerns. Να σας ενημερώσω λοιπόν για αυτά τα οποία εξέφρασαν ανησυχία οι βουλευτές για την ε, αποτίμηση πριν από την ε, εξυγίανση και υπάρχει ένα πρώτο ζήτημα εκεί πέρα. Μετά στην παράγραφο 5 οι εκφράσεις μπορεί να ισχύσει και όπου δι χρησιμοποιούνται. Αλλά τώρα έχουν έρθει οι προσκεκλημένοι μας, οπότε μπορώ να σταματήσω και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των βουλευτών, ξεκινώντας βεβαίω με τα μέλη τα, της ομάδας διαπραγμάτευσης της οδηγίας ε, τραπεζών. Δίνω τον λόγο στον κύριο Τορνέζε, τον Εμιλιάνο Τορνέζε, ο οποίος ε, είναι αρμόδιος για τα θέματα διαχείρισης κρίσεων και εξυγίανση. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, σας ευχαριστώ που μας ε, προσκαλέσατε στην συζήτηση των, του σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Εξυγένσης, δηλαδή της σχετική οδηγία και του μηχανισμού ε, Εξυγένσης. Πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα και αυτό φαίνεται από το ότι οι ειδικοί εργάζονται για τις τεχνικές αυτές προδιαγραφές εδώ και καιρό μαζί μας. Τα σχέδια αυτά ρυθμιστικών ε, τεχνικών προδιαγραφών, ενώ αφορούν και τα δύο το ζήτημα της αποτίμησης, ε, αφορούν δύο σημαντικά τμήματα της διαδικασίας. Το ένα αφορά το κομμάτι προ και μετά εξυγίανσης. Ε, Πρώτη εξυγείας λοιπόν η αποτίμηση έχει στόχο να ξεκαθαρίσει το πώς θα γίνει η αποτίμηση από τις αρχές ε, εξυγίανσης έτσι ώστε η τράπεζα να πληρεί τους όρους ε, για την εξυγένση ή για την διαγραφή κάποιων κεφαλαίων. Ο δεύτερος στόχος είναι βασικά να να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την δράση η οποία θα αναλυφθεί έτσι ο στόχος της εξυγίανσης να επιτευχθεί με το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η οδηγία απαιτεί η αποτίμηση αυτή να αναγνωρίζει πλήρως οποιασδήποτε ζημίε της τράπεζας ή ε, υποεξυγίανση και έτσι να γίνεται με τρόπο δίκαιο και ρεαλιστικό. Όσον αφορά λοιπόν το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προδιαγραφών, μιλάμε για το τι θα γίνει μετά την εξυγίανση και βεβαίως έχουμε την αρχή η οποία υπάρχει, η οποία είναι ότι κανείς πιστωτής δεν θα πρέπει να είναι σε χειρότερη θέση και ο στόχος είναι οι μέτοχοι και οι ψωτές ε, της ε, τράπεζας να μην έχουν χειρότερη μεταχείριση σε σχέση με το τι θα είχαν εάν η τράπεζα ακολουθούσε κανονικές διαδικασίες χρεοκοπίας. Οπότε, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, η εφαρμογή αυτής της ρήτρας είναι πάρα πολύ σημαντική για... στο πλαίσιο και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων για να μην επηρεάζονται τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία των μετόχων και των πιστωτών και για να προστατευτεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτή λοιπόν είναι οι δύο στόχοι των ρυθμιστικών τεχνικών προδιαγραφών ε, του πρώτου και του δεύτερου πακέτου. Όπως είπα, είναι ένα μάλλον τεχνικό και περίπλοκο ζήτημα. Ε, εμείς έχουμε συζητήσει τη συμμετοχή μας ως παρατηρητές ε, στις εργασίες Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Απαιτείται αρκετές αλλαγές στην διαδικασία, αλλά τελικά θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό όσον αφορά τα μέτρα επίπεδου 1 της οδηγίας ανακαμψής και εξήγησης τώρα τα εγκρίνουμε εσωτερικά στην Κομισιόν υπάρχουν κάποια σχόλια που έχουν γίνει από τις διάφορες υπηρεσίες μας οι μικρές αυτές αλλαγές δεν θα αλλάξουν την ουσία του σχέδιου αυτού όπως το παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και μπορώ να πω ήδη πως ε, ένα από αυτά τα ερωτήματα ξεκίνησε μια διαδικασία επανεξέτασης και πλέον προχωράμε σε διευκρινήσεις στο κείμενο. Σας ευχαριστώ. Ε, ποιο ζήτημα ήταν αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Να σας πω αμέσως. Αφορά το πώς οι αξιολογητές μπορούν να κάνουν την αποτίμηση. Στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής προτείναμε ένας ανεξάρτητος να μπορεί να κάνει πολλαπλές αποτιμήσεις ετέθη ένα ερώτημα από έναν βουλευτή που είπε πως θα ήταν καλό να έχουμε περισσότερους αξιολογητές κάτι το οποίο εξετάσαμε και θεωρούσαμε ότι καλό θα ήταν να αλλάξει το κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα πράγματι μοιάζει μια βελτίωση λέει ο πρόεδρος ωραία τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ και της Διαπραγματευτικής Ομάδας. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για τη μεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρμόζονται για ε, την αξιολόγηση που ζητείτε. Το RTS ε, συνιστά ένα σημαντικό βήμα πρόοδου ε, στις δράσεις εξηγίας πάντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε απόφαση για την εξηγήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από μία αξιολόγηση με τεχνικά στοιχεία ακριβώς για την δράση αυτή. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν για τις ε, συνθήκες ε, ε, για την εξυγίανση και επίσης το κατά πόσο τα μέσα εργαλεία κεφαλαίου και τα στοιχεία του παθητικού χρησιμοποιούνται στη μετατροπή. Ένας ανεξάρτητος αξιολογητής επιφορτίζεται με την αξιολόγηση και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να γίνει αυτό με μια προσωρινή αξιολόγηση από την ίδια την αρχή ε, εξηγένσης. Ε, θα πρέπει όμως πάντα αργότερα να ακολουθεί αξιολόγηση από ανεξάρτητο αξιολογητή. Η αξιολόγηση είναι κρίσιμη για την εξηγίαση. Ε, τροφοδοτείται και ε, αλληλεπιδρά με τις ε, ρευστές συνθήκες που επικρατούν όταν ένα ίδρυμα βρίσκεται σε δινή θέση. Και χρειάζεται τεχνική υποστήριξη για να αποφευθεί ο ηθικός κίνδυνος της θάλασσας, να μην επιβαρυνθεί όσο γίνεται ο φορολογούμενος και να σεβόμαστε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία αυτοί που θα πρέπει να χάνουν πρώτοι είναι οι μέτοχοι και οι ε, πιστωτές. Αυτό ε, αφορά επίσης ε, και περιπτώσεις τύπου κουρέματος και άλλων κεφαλαϊκών μέσων. Αυτό δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το νέο αγοραστή ή το νέο ιδιοκτήτη. Επίσης θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η ε, ε, κρατική υποστήριξη, η κρατική ενίσχυση. Άρα απαγορεύεται ε, ο αξιολογητής ή η αξιολόγηση να δέχεται ως ενδεχόμενο την κρατική ενίσχυση. Το ενεργητικό και το παθητικό θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση στοιχεία δίκαια, ασφαλή και ρεαλιστικά και με σύνεση. Ε, οι στόχοι ε, να επιτυχάνονται και η όλη αξία είναι ε, να χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζει το εργαλείο Bain και να συνεχίσει τη λειτουργία της η τράπεζα. Όταν όμως πρόκειται να πωλήσει θα πρέπει να αξιολογείται διαφορετικά. Η ε, τιμή πώληση βασίζεται στις ε, τιμές της αγοράς και μπορεί να έχει να κάνει και με ε, στοιχεία μη ρευστά. Η αλληπίδρυση με το πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης εμφανίζεται επίσης αντανακλάτες στο RTS έτσι ώστε όταν έχουμε NPLs ή άλλα στοιχεία ενεργητικού μεταφέρονται σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσίας ε, και η ενδεχόμενη αξία αυξάνεται ε, σε ένα μακροπρόθεσμο και μακροχρόνιο ορίζοντα. Ε, όταν γίνεται λοιπόν εξολόγηση πριν από την εξυγίανση, ο ανεξάρτητος αξιολογητής καλείται να εκτιμήσει και σεβόμενος τα δικαιώματα των μετόχων και των πιστωτών. και θα πρέπει να σέβεται την αρχή του να μην βρίσκεται κανείς πιστωτή σε ε, ε, χειρότερη μοίρα από τον άλλο no creditor wars off όπως συμβαίνει σε ε, κανονικές διαδικασίες αφαιρεγγιότητας και πτώχευσης. Επίσης υπάρχει και μία εκ των υστέρων αξιολόγηση που έρχεται να εκτιμήσει ε, κατά πόσο οι μέτοχοι και οι πιστωτές έχουν ε, υποστεί ε, μεγαλύτερες απώλειες από την εξυγίανση παρά αν είχε ακολουθηθεί μία κανονική διαδικασία πτώχευσης. σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποζημιωθούν από το Ταμείο Εξυγίανσης οι ελόγω μέτοχοι, οι πιστωτές. Αυτό όμω διαφέρει εκ των υστέρων αξιολόγηση από την εκ των προτέρων γιατί βασίζεται σε ένα υποθετικό σενάριο και όχι στην πραγματική ε, ε, συναλλαγή και στον πραγματικό υπολογισμό. Η υποθετική ε, αποζημίωση βασίζεται και υπολογίζεται με βάση το κείμενο πτωχευτικό δίκαιο και την πρακτική που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον συντονιστή μας για την οδηγία, τον ε, κύριο Χόκμαρκ. Ευχαριστώ. Ε, ο εισαγητής ο κύριος Χόκμαρκ, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Τραπεζικής Αρχής και, ε, την, ε, και για την παρουσίασή σας. Έχουμε κάποιες ανησυχίες λόγω του μεγέθους αυτής της αλλαγής, όπως αντιλαμβάνομαι. Το ζήτημα είναι αν θα πετύχουμε μεγαλύτερο επίπεδο βεβαιότητας εάν θα έχετε και τη δυνατότητα να ε, έχετε κάποιο περιθώριο της ε, δικής σας διακριτικής ευχέρειας στα θέματα της εξυγίανσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αξιολόγησε τα σχετικά θέματα αναφέρατε ένα σημείο για το αν θα είναι ε, Σαλ ή Μέη η διάταξη. Νομίζω στο άρθρο 8 της επισκόπησης ε, αναφέρεται αυτό. Και επίσης τι μπορεί να γίνει για να διαλυθεί περισσότερο η ασάφεια και να μην χαθούν ευκαιρίες όταν ε, γίνεται η προσπάθεια εξυγένσης. Πόσο περισσότερα μπορούν να επιτευχθούν σε ένα πρόγραμμα εξυγίανση σε σχέση με τις επιμέρους τράπεζες. διότι πολλά νομίζω θα μπορούσαν να αποσαφενιστούν εκ των προτέρων στο πρόγραμμα εξυγίανσής σας. Εξαρτάται σε ποια φάση της βρίσκεται η τράπεζα όταν ξεκινά η εξυγίανση. Τι μορφή έχει αγορά, πώς είναι τα πράγματα. Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα. Τι μπορεί να κάνει για αυτά η Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Είναι και θεμητές και εύστοχες και αυτός είναι και ο λόγος που συζητούνται αυτά τα τεχνικά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή εδώ και κάποιο καιρό. Έχουμε τον στόχο της νομικής σαφήνειας, της νομικής ε, βεβαιότητας και γι' αυτό η αποτίμηση είναι περισσότερο τέχνη παρά ακριβής επιστήμη. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο να εκφραστεί με σαφείς αρχές και όρους. Η αρχή προσπάθησε και νομίζω αν θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε την απάντησή μου η έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και όταν αναφέρεστε στο Σάλ ή το Μέι Αυτή την ανησυχία την αναφέραμε και εμείς. Δεν θέλαμε να περιορίσουμε πάρα πολύ τη διακριτική ευχέρεια των αξιολογητών για να μπορούν να είναι ως το δυνατόν πιο ελεύθεροι στην αξιολόγησή τους. Στο δεύτερο σετ των προτύπων ε, αναφέρεται και πάλι το ΣΑΛ και το ΜΕΙ και καλό είναι να μην κάνουμε πιο αυστηρά τα κριτήρια αλλά να μπορεί ο αξιολογητής να τα χρησιμοποιήσει κάπως ελεύθερα εφόσον τεκμηριώνει τη χρήση τους και αιτιολογείται αυτό στην έκθεση αποτίμησης. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε όσο σαφείς όσο επιτρέπεται σε μια τέτοια προσπάθεια. Κάτι τέτοιο πρέπει να το πετυχαίνει, επιτυγχάνει το νομικό κείμενο, αλλά πρέπει να δίνουμε και την ευκαιρία στον αξιολογητή. και να μπορεί και ο άλλος αξιολογητής να το λάβει υπόψη του πριν καταλήξει την τελική αποτίμηση. Αυτή ήταν λίγο πολύ η δυσκολία μας. Ναι, απλώς να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε για το πόσο περισσότερο μπορούμε να πετύχουμε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης. Πολύ καλή παρατήρηση. Διότι πάει στο της ετοιμότητας για εξυγίανση και γιατί χρειάζονται υποτιμήσεις. Οι αποτιμήσεις βασίζονται σε συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων και τα σύνολα δεδομένων απαιτούν δεδομένα. Αυτό είναι μέρος της ετήσιας διαδικασίας συλλογής δεδομένων και της δοκιμασίας της αντοχής των τραπεζών και ούτω καθεξής. Είναι μέρος λοιπόν όλης αυτής της διαδικασίας των ρυθμιστικών τεχνητών, τεχνικών προτύπων. Αυτήν την ε, προσέγγιση μπορούν να την ακολουθήσουν οι αποτιμητές Τώρα ε, αυτό το κάνουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι αποτιμητές ε, κοιτάζουν τη δυνατότητα των τραπεζών να προσφέρουν ποιοτικά δεδομένα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε. Περβάνς Μπερές. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας δεν καθορίζεται από τις ανάγκες της πραγματικότητας ή τη βούληση του νομοθέτη, όμως πολλά έχουν γίνει έκτοτε και είναι δύσκολο να κοιτάξουμε τα RTS χωρίς να λάβουμε υπόψη τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είχαμε μια επιτυχή εξυγίανση, αλλά να σκεφτούμε το παράδειγμα της Banco Popular. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία, ιδίως το θέμα της αποτίμησης ακριβώς. Όλο το θέμα έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα από την αρχή, αλλά λαμβάνουμε διαρκώς επιστολές που μας λένε ότι το Banco Popular είχε μηδενική αξία αρχικά και τώρα είναι πολύ ψηλά στην αγορά. Η συγκεκριμένη μου ερώτηση λοιπόν είναι εάν αυτά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα είχαν ισχύσει, είχαν εφαρμοστεί θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα της περίπτωσης του, της Banco Popular και αν ναι, πώς θα είχε επηρεαστεί όλη τη δικασία. Δεν ξέρω αν είμαστε κυκλισμένοι των θυρών και μπορείτε να μιλήσετε τελείω ανοιχτά, αλλά ελπίζω και πάλι να μπορείτε να απαντήσετε ελεύθερα στην ερώτηση. Και η δεύτερη έχει να κάνει με την αποτίμηση και το πόσο αυτή ε, αφορά την εμπιστοσύνη και την ε, αξία που της δίνεται. Όχι μόνο δηλαδή η αγορά να λαμβάνει υπόψη και να δέχεται την αποτίμηση, αλλά και η διαφάνεια και η μεθοδολογία της διαδικασίας. Εάν εγκριθούν αυτά τα τεχνικά πρότυπα, θα κινηθούμε στη σωστή κατεύθυνση. Εύκολη ερώτηση, θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Είναι ουσιαστική ε, ερώτηση. Αλλά βεβαίως θα την συνέδεα τη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι μια απόφαση εξυγίανσης ε, που ελήφθη από μια ανεξάρτητη αρχή όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας ε, που έκανε την αξιολόγηση αυτή με την έγκριση της Κομισιόν. σε αυτή την περίπτωση εξηγένση όπω οποιαδήποτε άλλη θα έλεγα πως ε, το πρώτο σχέδιο των ρυθμιστικών τεχνικών προδιαγραφών είναι δημόσιο εδώ και καιρό. Υπήρξε διαβούλευση. Έχει εγκριθεί επισήμω ε, ε, από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή το Μάιο 2017 και βέβαια οι αλλαγέ αυτές δεν είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να αλλάζουν την ουσία της, εκτός από τις ε, διευκρινήσεις που δόθηκαν. Αλλά και πάλι δεν θα επηρεάζει την ουσία του αρχικού κειμένου. Αλλά αναφερθήκατε, σωστά, στην ανάγκη να εγκριθεί ε, αυτό το κείμενο του σώμα των δυνατών, αλλά και στις ανησυχίες ε, για το πόσο μπορούμε να έχουμε νομική σαφήνεια και βεβαιότητα σε τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό χρειάστηκε λίγος χρόνος αν μπορώ να αποκαλύψω κάτι, το κείμενο ε, εσωτερικά το επεξεργαστήκαμε πάρα πολύ από το πρώτο σχέδιο. Οπότε χρειάστηκε χρόνος γιατί είναι περίπλοκα τεχνικά ζητήματα και να λάβουν υπόψη ότι βεβαίως το πώς εφαρμόζονται τα λογιστικά πρότυπα δεν ε, είναι πάντα το ίδιο για όλα τα κράτη-μέλη και τις αρχές. Οπότε τώρα που είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, τώρα που εγκρίθηκε τελική απόφαση και είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε, ε, είναι κάτι το πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Συγγνώμη γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε πλήρως ή να σχολιάσετε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις από τεχνική σκοπιά εάν οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές ήταν ήδη νόμους ε, τεχνικά μιλώντας θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι ε, διαφορετικό διαδικαστικά ή η διαδικασία η οποία εγκρίθηκε είναι ακριβώς η ίδια η οποία περιέχεται στις ε, ρυθμιστικές τεχνικές προδιαγραφές και δεν θα είχε αλλάξει τίποτα. Τώρα το αν ε, αυτό το οποίο συνέβη ήταν σωστό, αν ήταν υπερτιμημένο ή υποτιμημένο, δεν είναι τώρα η στιγμή να απαντηθεί, αλλά το κομμάτι αυτό τη ερώτηση νομίζω αξίζει να απαντηθεί. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, δυστυχώ. δεν μπορώ να απαντήσω για έναν απλό λόγο, γιατί το επίπεδο 1 της οδηγίας ε, απαιτεί αξιολόγηση να γίνει από ανεξάρτητο αξιολογητή. Το γεγονός ότι οι τεχνικέ αυτέ προδιαγραφέ ήταν δημόσιε, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέτρο σύγκριση. Αλλά βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο θα αξιολογήσει μόνο ο αποτιμητή. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι σε θέση να πω το εάν ε, θα ήταν ε, διαφορετική η απόφαση, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι οι ρυθμιστικές τεχνικές αυτές τις αντικατοπτρίζουν τις πρακτικές αποτίμησης και οπότε θα έλεγα δεν θα άλλαζε η ε, διαφορετική θέση. Γιατί? Γιατί ήταν ε, δημόσιες και δεν θα άλλαζε ο τρόπος ε, διεξαγωγής αυτών των περιπτώσεων. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Μπέρες και δεν ακούγεται. I'm sorry, I didn't... Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Όχι, έλεγα, ακούγοντάς σας, λέτε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές ακολουθούν τη συνήθη πρακτική. Και ποια είναι η συνήθις πρακτική. Γιατί λέτε ότι στο παρελθόν άλλαζαν πολύ συχνά ε, τα πράγματα λόγω της πρακτικής διαφορετικής που ακολουθούσαν εκάστοτε. Οπότε δεν είναι τόσο σαφή για τη συνήθη πρακτική και για τη διαφάνεια δεν απαντήσατε. Αναφέρω όμως στο παρελθόν, στην προηγούμενη περίοδο, μέχρι το 2015. Το κείμενο του 2017, του Μαΐου συγκεκριμένα, ε, είναι αρκετά ε, σταθερό και εγκρίθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και είναι και αναφορά για την αγορά. Αλλά όταν ρωτούσαν πότε θα εγκριθούν αυτές οι προδιαγραφές, τους παραπέμπουμε στην έγκριση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Ξέρουν δηλαδή οι φορείς της αγοράς που να κινηθούν σε ποιο πλαίσιο. Υπάρχουν έγγραφα από τους διάφορους οργανισμούς αρμόδιοι. Για τη διαφάνεια μπορείτε σας παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτησή σας γιατί εστίασα περισσότερο στα τεχνικά. Αυτό το θέμα της αποτίμησης, εκτίμησης έχει να κάνει ε, ουσιαστικά με την εμπιστοσύνη και πάνω από τη μεθοδολογία έχει σημασία το κοινό και οι ενεχόμενοι να έχουν μια σαφή εικόνα για το πώς εφαρμόζεται και με πόσο διαφανής είναι όλη η διαδικασία, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση αυτή. Έχει υπάρξει καμία βελτίωση στον τομέα αυτό. Αποδίδεται καμία σημασία σε αυτά τα θέματα της διαφάνειας. Βεβαίως είναι βασική η διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Έχουμε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές που θέλουμε το συντομότερο να εγκριθούν και βασίζονται σε αρχές. Ποιες είναι αυτές. Είναι αρχές που θα πρέπει να ακολουθούν και να τηρούν όλοι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές, αλλά είναι απόκειται και στον εκάστοτε ανεξάρτητο ε, αξιολογητή να τηρεί τους κανόνες ο ίδιος. Η ίδια η διαδικασία αυτή της εκτίμησης, αποτίμησης, αξιολόγησης δεν ε, οφείλει να δημοσιεύεται βάσει ε, του μέτρου του πρώτου επίπεδου και είναι και πάρα πολύ τεχνική και μετά ακολουθεί η απόφαση για την εξυγίανση. Είναι κάποια στοιχεία που μπορούν να δημοσιεύονται ας πούμε, οι αρχές που θα πρέπει να τηρεί και να υιοθετεί ο ανεξάρτητος εκτιμητής και μετά υπάρχει το τελικό προϊόν που είναι ειδικό για την κάθε περίπτωση και θα πρέπει να εκτιμάται ε, αν υπάρχουν κάποια νομικά ζητήματα και κάποιος έλεγχος. Στο επίπεδο 1 όμως, και δεν είναι κακό αυτό, δεν οφείλει να δημοσιεύεται όλη αυτή η διαδικασία για το ευρύ κοινό. Ευχαριστώ. Ο Φίλιπ Λάμπερτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως, η αποτιμήση είναι μια τεχνική διαδικασία. Αλλά, τι σημαίνει αυτό ότι είναι καθοριστικό ότι ανάλογα με το πόσο θα εκτιμήσεις την αξία ε, θα την πληρώσει ο φορολογούμενος ή όχι. Δηλαδή κάποιος ε, θα χάσει χρήματα με βάση την εκτίμηση στην οποία θα καταλήξει. Εκπλήσουμε λίγο από την αντίφαση των λεγόμενων σας. Λέτε ότι η οχι δηλαδη καποιο θα χασει χρηματα με βαση την εκτιμηση είναι τέχνη και συμφωνώ. Αλλά πώς μπορείτε να λέτε μετά ότι είναι προαιρετικό να προτείνει κάποιος τιμές. Δηλαδή είτε είναι επιστήμη και η εξίσωση βγάζει ένα αποτέλεσμα είτε είναι τέχνη και πρέπει να έχεις έτσι διάφορες επιλογές να επιλέξεις. Πώς το ερμηνεύω εγώ. Όταν λέτε ε, ότι είναι προαιρετικό να δίνει κανείς κάποια τάξη μεγέθους, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει εκεί. Η αρχή που είναι αρμόδια για την εξυγίανση θα βγει να πει στον αξιολογητή θέλω να μου φέρεις ε, αριθμό, ποσό. Ε, κάνοντας αυτό όμως μεταφέρεται η ευθύνη της απόφασης από την αρχή που είναι αρμόδια για την εξυγίαση στον εκτιμητή και θα βγει και θα ανοίξει τα σχήρα της και θα πει ότι εγώ δεν φταίω. Αυτό μου είπε ο αξιολογητής ότι αξίζει, πουλάω την τράπεζα και δεν είναι δική μου ευθύνη. Ενώ ο νομοθέτης έχει αποφασίσει την ευθύνη να τη φέρει η αρχή που είναι αρμόδια για την εξυγίαση. Και προσωπικά, ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο εξακολουθείτε να αρνείστε να είναι κανόνας και να ισχύει η αρχή ότι οι αξιολογητές φέρουν κάποιες προτάσεις σε τάξη μεγέθους. 4,9 δις ας πούμε ε, με 4,95 δις. Μπορεί να είναι αυτό το περιθώριο πολύ στενό, δεν χρειάζεται να εύρει. Γιατί δεν κάνετε αυτή τη ρύθμιση. Και οι αξίες μετά θα βασίζονται σε κάποιες παραδοχές που γίνονται και όχι σε ε, έλλειψη πληροφόρησης. Ε, ε, αν είμαι εγώ λοιπόν ο εκτιμητής, εγώ τι θα κάνω, θα σας φέρω μία τάξη μεγέθους και θα αποφασίσετε εσείς ποια αξία θα δεχθείτε. Και πάλι αυτό είναι η ευθύνη, είναι ευθύνη μάλλον, της αρμόδιας για την εξυγίανση αρχής να, να πάρει την απόφαση να κινηθεί Προ το φορολογούμενο. Δηλαδή, ε, έχει μια τιμή. Ε, παίρνω τη τιμή, τη λαμβάνω υπόψη, ε, αυτό το περιθώριο που μου δίνεται, για να προστατεύσω το φορολογούμενο όμως, παίρνω τις αποφάσεις... Δεν ξέρω, μπορεί να με θεωρείτε υπερευαίσθητο, αλλά είδα τι έγινε πρόσφατα στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά κυρίως στην Ιταλία. Και τι εννοώ, ότι όταν αφήνεται πολύ χαλαρά όλα αυτά τα πράγματα, ε, χωράνε διάφορες ερμηνείες οι οποίε τελικά δεν είναι ευνοϊκέ για το φορολογούμενο. Είδαμε τι απαντήσει τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, δεν μα πείθουν ακριβώ. Και πέρα από το γεγονό ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα ε, ε, κάποια τάξη μεγέθους, όχι ό, όταν αυτό ενδείκνεται. Αυτό ενδείκνεται πάντα και όταν χρειάζονται περισσότερες εκτιμήσεις να γίνονται από ανεξάρτητους εκτιμητές, όχι τον ίδιο, περισσότερους του ενός. Πώς ερμηνεύετε τους κανόνες επιστοτές μπορούν ε, οι πιστωτές ε, να ισχυριστούν ε, ότι οι απαιτήσει τους πρέπει να ικανοποιηθούν γιατί δεν είναι τελείως αφαιρέγγια η τράπεζα ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να εκποιηθούν και να αποπληρωθεί το χρέος. Κάποια άλλα τεχνικά που θα πρέπει να ισχύουν για όλους και όχι αναπερίπτωση. Εμείς ως Επιτροπή που θέλουμε να ακούσουμε και να λάβουμε ε, υπόψη αυτά που λέτε. Θέλουμε να μας λάβετε και εσείς υπόψη σε αυτά που λέμε. Ευχαριστώ. Βεβαίω δεν είναι μόνο οι φορολογούμενοι, αλλά έχουμε και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Γι' αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία η αποτίμηση. Ναι, ναι, και πάλι, αλλά είναι και πάλι ιδιοκτησία των φορολογουμένων. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούμε λεφτά των φορολογουμένων, αφαιρούμε ιδιοκτησία των φορολογουμένων. Συγγνώμη. Μα ναι, είναι βέβαιες και έχουμε μπλε, έχεις εμπλακεί σε μια κατάσταση στην οποία μπορούσε να μην είχες μπλέξει. Αλλά ο καταναλωτής δεν είναι, ο φορολογούμενος δεν έχει επιλογή γιατί ο κάθε φορολογούμενος εμπλέκεται από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Δεν εμπλέκονται όλοι όμως ε, σε μια συγκεκριμένη τράπεζα και όταν πας σε μια τράπεζα πάντα έχεις την επιλογή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, δεν ε, καταλάβατε μάλλον το τι είπα. Είπα ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που επηρεάζονται από την αποτίμηση. Και πιθανώς να μην επηρεάζεται ο φορολογούμενος, αλλά μια αποτίμηση μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη και να δημιουργήσει συζητήσεις. Γι' αυτό υπάρχει το θέμα της διαφάνειας που Λοιπόν, ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος. Ναι, ναι να απαντήσω εγώ και μετά και ο συναδελφός μου για το πρώτο θέμα το οποίο θίξατε. Ίσως υπάρχει κάποια ασάφεια και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αρχή εξυγίανσης θα λάβει την ε, τελική απόφαση, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το ευρώ. Αλλά πρέπει να μιλάμε για δύο αποτιμήσεις. Η πρώτη αφορά ακριβώς το εάν μία τράπεζα ε, χρεοκοπεί ή όχι και εκεί πέρα χρειαζόμαστε απόλυτη βεβαιότητα και μετά περνάμε στο δεύτερο ερώτημα και εκεί πέρα χρειάζεται ένα εύρος, ένα φάσμα και εκεί πέρα έχετε δίκιο ο ανεξάρτητος αξιολογητής θα κάνει αυτή την πρόταση αλλά θα αποφασίσει μετά η οχι και εκει περα χρειαζομαστε απολυτη βεβαιοτητα και μετα περναμε στο δευτερο ερωτημα και εκει περα χρειαζεται ενα σε ενα φασμα και εκει περα εχετε δικιο ο ανεξαρτητος αξιολογητης θα κανει αυτη την προταση αλλα θα αποφασισει μετα η αρχη της εξυγίανσης με βάση το φάσμα ποιο είναι το καλύτερο, ακόμα και για την πρώτη αξιολόγηση, αποτίμηση. Πώς μπορείτε να είστε βέβαιοι όταν βασίζεται και η αποτίμηση ένα σε υποθέσεις πάντα. Έχουμε βεβαιότητα όταν έχουμε μία αποτίμηση και όχι ένα φάσμα. μικροφώνου Είναι καλύτερο να έχουμε ένα φάσμα για την αποτίμηση, αλλά θα δώσω τον λόγο στην ΑΛΦΑ από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ευχαριστώ. Θέσατε κάποια καλά ερωτήματα. Νομίζαμε ότι τα απαντήσαμε επαρκώ. Να, να απαντήσω πάλι για το εύρος αυτό της αποτίμησης σε σχέση με την σημειακή εκτίμηση. Είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή τα μοντέλα δίνουν ε, ένα φάσμα αποτίμησης και οποιοδήποτε σημείο εντός ε, αυτού του φάσματος βεβαίως εξαρτάται από τις πιθανότητες ε, τις αιρέσης που υπάρχουν και τις ελλείψεις. Και βεβαίως ο Εμιλιάνο είπε ότι έχουμε εξοδέψει πολύ χρόνο συντάσσοντας αυτές τις ρυθμιστικές τεχνικές προδιαγραφές και ακριβώς αυτό το θέμα συζητούσαμε. Δεν θέλουμε να μεταφέρουμε την ευθύνη. Η ευθύνη, όπως είπατε, είναι της αρχής εξυγίανσης. Η αβεβαιότητα είναι μια δυσκολία της διαδικασίας. Ειδικά στην προσωρινή αποτίμηση, εκεί όπου λέμε εάν χρεοκοπεί ή όχι ένα ε, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Και εκεί ακριβώς ε, ένα διάλειμμα το οποίο δεν θα, ένα διάστημα το οποίο δεν θα ήταν πολύ ακριβές προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητα για το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εάν επιλέξουμε μία επιλογή σε σχέση με μία άλλη. Γι' αυτό ακριβώς εμείς εάν ε, ήμασταν η αρχή εξηγένσης θα ζητούσαμε την καλύτερη ακριβή εκτίμηση από ολόκληρο το φάσμα. αυτό ακριβώς. Ε, αυτό σημαίνει δηλαδή η σημειακή εκτίμηση και με βάση αυτό λαμβάνεται η απόφαση. Για τις λοιπές αποτιμήσεις, μου επιτρέπετε να τελειώσω. Υπάρχουν σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Το ότι υπάρχει αποτίμηση 3. Το ότι υπάρχει αποζημίωση. Αυτό φορά αυτό το οποίο είπατε για το ότι οι αξίες δεν αντικατοπτρίζονται σωστά ή τη σχετική αβεβαιότητα ε, το αν αντικατοπτρίζονται σωστά από την αποτίμηση. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να γίνει αποτίμηση ε, περισσότερες φορές με πλήρεις πληροφορίες και να αξιολογήσουμε μετά το τι έχει συμβεί στην αξία. Τελικά, το θέμα είναι ότι η εκτίμηση πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία. Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω, γιατί αν είναι πιο κάτω, τότε ουσιαστικά επιδοτούμε αυτόν ο οποίος θα λάβει αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού μετά την εξηγένση. Γι' αυτό θεωρούμε τελικά ότι αυτές οι ρυθμιστικές τεχνικές προδιαγραφές ε, και το επίπεδο είναι ουσιαστικά έχουν τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Και για τα άλλα δύο σημεία... Α, να σταματήσω. Για τα άλλα δύο σημεία, για το θέμα της δυνατότητας ε, να έχουμε πάνω από έναν ε, ανεξάρτητο εκτιμητή. Έχουμε κάνει αυτή την διευκρίνηση. Έχουμε πει ποια είναι η μόνη έλλειψη υπάρχει, δηλαδή χρόνος και πολυπλοκότητα της διαδικασίας και όσον αφορά τον ε, ορίζοντα, τον κοινό ορίζοντα εκποίησης, είναι μια ιδέα δύσκολη στο να υλοποιηθεί, να σκεφτούμε και την διαφορά μεταξύ των διαφόρων στοιχείων ε, ενεργητικού που αξιολογούνται. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρούμε ένα ελάχιστο μήνυμο που θα επαρκεί για όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό δεν το ακολουθήσαμε. Ευχαριστούμε, Φίλιπ. Ναι. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει η περίπτωση του Μπάνκου Παπουλάρ στα δικαστήρια. Εάν κερδίσουν, τι θα γίνει με την αποτίμηση όμως, το βάρος θα το έχουν εκείνοι. Βεβαίως, η κάθε αξιολόγηση και το κάθε σημείο που αξιολογείται σε κάθε στιγμή έχει και ένα κάβεατ από πίσω. Είναι μια προειδοποίηση, υπάρχει ένα περιθώριο λάθος. Όμως το, η αποτίμηση θα πρέπει να λέει το φάσμα του καλύτερου και του χειρότερου σενάριου είναι αυτό Υπάρχουν και κάποιες ικαεσίες που συνοδεύουν όλα αυτά τα σενάρια και οι αρχές πρέπει να αποφασίζουν ποια αξία και τιμή θα πιστέψουν. Καταλαβαίνω ότι θέλετε την κάλυψη της αρχής της εξυγένσης, γιατί θα λένε δεν ξέραμε τι ψαλίδα υπάρχει, εμείς πήραμε μόνο τους αριθμούς. Και μπορείτε να κρυφτείτε πίσω αυτούς τους αριθμούς και να πείτε ότι δεν είχαμε τιμή. Όμως είναι καλύτερα να πάρετε την ψαλίδα και από την πρώτη αποτίμηση και να υπάρχει αυτό το φάσμα δυνατοτήτων. Γιατί να μην δώσει αποτιμητή όλο τον ντοσιέ και βάσει όλη τη δουλειά, όλων των πληροφοριών που είχε, αυτό το, το, το φάσμα, αυτή την ψαλίδα μπορούμε να καλύψουμε. Και σας συνιστούμε να πάρετε αυτή την αξία ή αυτή την τιμή ή την άλλη, αλλά είναι συμβουλή. Δεν είναι ακριβώς καταρτισμένος αριθμός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ε, να απαντήσω γρήγορα σε αυτό. Νομίζω το επιχείρημά σας που έχει να κάνει με τη μεταφορά των ευθυνών από την αρχή της εξυγίανσης στον ανεξάρτητο αξιολογητή, αυτό δεν στέκει. δεν είναι θέμα ψαλίδας ή ποσοστίων μονάδων. Η αποτίμηση συνήθως δίνει ως συμπέρασμα ότι είναι προσωρινή. Η προσωρινή προσυπογράφεται από την αρχή εξυγένσης. Συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε, αλλά ό,τι και αν πει η ανεξάρτητη αποτίμηση είναι μια συμβολή στη λήψη απόφασης από την αρχή εξυγένσης. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι η αποτίμηση Ναι, αλλά πώς θα διδράσουν τα δικαστήρια. Η αρχή εξυγένση θα πει είχαμε έναν αριθμό μόνο βάσει το οποίο μπορούσαμε να, να αποφασίσουμε και βάσει αυτού του αριθμού είπαμε το fail likely to fail. Μπορεί να πτωχεύσει, πτωχεύει. Δηλαδή οι αποτιμητές είχαν διάφορους αριθμούς στα χέρια τους. Ε, τους ζητήσαμε κάποιον μας έδωσαν αυτό, ήταν, ήταν άλλος, μπορεί να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του fail ή likely to fail. Οπότε, ποιο αποφασίζει τελικά αυτό ο ένα αριθμό ποιο θα είναι. Ναι, ίσω ένα τελευταίο πράγμα. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η αποτίμηση ε, του αποτυγχάνει, που πτωχεύει ή μπορεί να πτωχεύσει είναι κάτι που μπορεί να το αποφασίσει ο επόπτης. Εδώ μιλάμε για ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αποτίμηση, τέλο πάντων την ε, πρώτη αποτίμηση τη αρχής εξυγίανση. Ο επόπτης που επιβλέπει την τράπεζα θα ε, λάβει την τελική απόφαση για το αν η τράπεζα πτωχεύει ή όχι. Είναι νομίζω μικρό το περιθώριο να υπάρχει τέτοια ε, εκμετάλλευση αυτού του θέματος, διότι υπάρχουν δύο αρμόδιες αρχές, και η εποπτική και η αρχή εξυγένσης, που μπορούν να αποφανθούν αυτό μας δίνει κάποια αυτοπεποίθηση για την αποτίμηση 1. Ωραία. Γκούναρ, θες κάτι? Ναι, μια πολύ σύντομη σκέψη γιατί θα το ξαναδούμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν συζητάμε τις διαφορετικές εναλλακτικέ, έχουμε λίγο την εντύπωση ότι θα έχουμε την τέλεια αποτίμηση η οποία όμως εξορισμού δεν πάβει να είναι αποτίμηση χωρίς καμία βεβαιότητα σε καμία κατάσταση και σε καμία περίπτωση. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως το τραβάμε λίγο από τα μαλλιά. Δεν μπορούμε να βρούμε το τέλειο, την τέλεια λύση. Και είναι λογικέ οι απάντησει του, οι ερωτήσει του Φιλίπ, αλλά δεν είμαι βέβαιο ότι εδώ μπορούν να επιληθούν όλα αυτά. σω η Επιτροπή να μπορεί να το σκεφτεί λίγο παραπάνω. Ωραία. Άλλα σχόλια. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Γκούναρ, έχεις κάτι να προσθέσεις. Αν μπορούμε να μάθουμε τίποτα για τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά απαντήθηκε. Η Επιτροπή. Πρέπει να το δουλέψει. Αναμένουμε το τελικό κείμενο της Επιτροπής. Βρίσκω ότι είναι αρκετά λογικό και βρίσκω και λογικά αυτά που είπατε για τη δυνατότητα πολλαπλών αποτιμήσεων. Είναι σαφής βελτίωση, είναι θεμητή η συζήτηση για την ε, συγκεκριμένη υπόθεση που θα πάρει την πορεία της αλλά δίνει και την αφορμή να συζητήσουμε για το RTS. Μην τα μπερδεύουμε βεβαίω. Το Ευρωκοινοβούλιο αναλύει με προσοχή τις επιμέρους υποθέσεις αλλά με τον ίδιο τρόπο θα κοιτάξουμε να αποτιμήσουμε και σωστά και την τελική πρόταση της Επιτροπής για την αποτίμηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την EBA και την Επιτροπή για τη συνεισφορά της στην ε, διαδικασία αυτή ελέγχου. Meeting is closed. You would like to say something, please? Just a reflection which was coming now, uh, which address uh, Θέλετε να πείτε κάτι, είναι ένα στοχασμό που μπορεί να αποσαφηνίσει το όλο θέμα. Ότι η αποτίμηση μπορεί να γίνει από πολλούς αποτιμητές. Είναι γεγονός. Και αυτό μπορεί να δίνει τη λύση. Εάν ζητηθεί αποτίμηση δύο αποτιμητών, δεν θα υπάρχει απλώ ε, το φάσμα αυτό που λέτε, αλλά δύο διαφορετικέ αποτιμήσει. Οπότε η αρχή, εξηγένση αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη. Άρα με την αποσαφήνιση που μπορεί να προκύψει για άλλους λόγους, ίσως να λύνουμε το πρόβλημα. Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα βελτίωσης. Ναι, Γκούναρ, παρατείνουμε τις συνεδρίες με φιλοσοφικά ζητήματα. Πολύ συχνά η τιμή θα είναι διαφορετική έτσι κι αλλιώς. Είναι σαν να προσπαθεί η γάτα να πιάσει την ουρά της και να τρέχει γύρω-γύρω. Όταν, είναι εύκο... όταν επιτύχει η εξυγίανση θα κοιτάνε όλοι τις αποτιμήσεις των τελευταίων ημερών και θα θεωρούν αυτές υπεύθυνες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να φιλοσοφούμε για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Λήξη. Η επόμενη 6 Νοεμβρίου 3 με 6.